Καλησπέρα. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Συνεχίζεται μάλλον η συνεδρίασή μας. Κυρίες και κύριοι, Έχετε τα πρακτικά, υπάρχουν ενστάσεις παρακαλώ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά.